Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Έχουμε τις επεξηγήσεις ψήφου τώρα. Με πρώτο θέμα... Το πρώτο θέμα λοιπόν έλεγα είναι η έκθεση Κοβάτσε. 71η Σύνοδο τη Γενική Συνέλευση των Αμένων Εθνών. Πρώτο ομιλητή. Κύριος